Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για το HIV AIDS. Ο Επίτροπος Κάτι έχει το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο ζουν και συμβιώνουν με τον HIV AIDS εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση αυτής της ασθένειας, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε να εξαλείψουμε την επιδημία μέχρι το 2030, θα πρέπει να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Παρακαλώ πολύ, Πρόεδρε. αδελφοί, όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή, σα, παρακαλώ το συντομότερο δυνατόν και εφόσον είναι δυνατόν, ε, χωρί φασαρία, να βγείτε από την αίθουσα. Και αυτό ισχύει και για εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Herr Kollege, sagenhaft. Herr Gualtieri, Herr Gualtieri, Tajani, kannst du ε, Ταγιάννη, πες τον Γκουαλτιέρη να φύγει. Και ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε στην εξάλληψη της επιτιμίας του AIDS μέχρι το 2030, θα πρέπει να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, για να προλάβουμε τη διάδοσή του, να δώσουμε σε όλους την δυνατότητα μιας πρόορης διάγνωσης και να χορηγήσουμε την επαρκή θεραπεία σε όλους όσους τη χρειάζονται. Η Κομισιόν καλωσορίζει την συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για το ε, HIV-AIDS που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη. Στηρίζουμε την προσπάθεια μιας γρήγορης ανταπόκρισης ε, και προσήλωσης ε, το AIDS εξακολουθεί να επηρεάζει πολύ την υποσαχάρη Αφρική. Δύο στους ε, τρει που ε, μολύνονται από το ε, ε, AIDS βρίσκονται εκεί. Εδώ επίσης στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη, ε, οι μολύνσεις του από AIDS αυξάνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο για την εξάλληψη αυτής της επιδημίας στη γειτονιά μας και σε άλλες χώρες του κόσμου με αλληλεγγύη και πρόσθετη βοήθεια σε αυτές τις ε, χώρες που τη χρειάζονται περισσότερο. Τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα κυρίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοχετεύει την βοήθειά της στην ε, πρόληψη και τη θεραπεία του AIDS μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου για την φυματίωση, την ε, μαλάρια και την ανοσία δηλαδή για το AIDS. Ε, με 8 εκατομμύρια άτομα με αυτά τα χρήματα παίρνουν θεραπεία τα 50% των όλων των πόρων που δίνουν, ε, δίνονται στον κόσμο, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, είναι βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Και άλλα 470 εκατομμύρια προβλέπονται για την περίοδο 2017-2019 από τον προπολογισμό μας. Και αυτό θα το ε, προτείνουμε το, στην Σύνοδο των Δωρητών τον Νοέμβριο. Πέρσι αλλάξαμε την ε, προσέγγιση μας η οποία έγινε πια πιο ε, σφαιρική που προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες τόσο για το AIDS όσο και για άλλες ε, ασθένειες θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που πλήττονται περισσότερο να βελτιώσουν τις υγειονομικές συνθήκες και την ποιότητα του ύδατος. Αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια. Η χρηματοδότηση ιδιαίτερα σε χώρες μεσαίων εισοδημάτων θα πρέπει να αυξηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πρόοδο. Ε, εξαλείψαμε στην ε, πράξη τη μετάδοση από τις γυναίκες στα παιδιά και την έκθεση λοιπόν των παιδιών στον ιό του AIDS. Η, τα νέα κρούσματα μειώνονται. Η κάλυψη με θεραπεία είναι υψηλή. Όμως έχουμε και σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον πάνω από 300.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστούν θεραπεία καθόλου το αγωγή, δηλαδή καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους. 30.000 άτομα μολύνονται κάθε χρόνο, ακόμα και σήμερα. Ε, μπορεί να προληφθούν. Έχει το, το AIDS έχει κοστίσει εκατομμύρια ευρώ και κοστίζει. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την κοινωνία των πολιτών προσπαθεί να βελτιώσει τα διαγνωστικά τεστ ε, και να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγωγή και τη θεραπεία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ιδιαίτερα την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, όπου εκεί τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται. Και πάλι θα είναι μια συλλογική προσπάθεια. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας σε όλες αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μπουσόη τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρετίζω την παρουσία του κυρίου Επιτρόπου εδώ στην σύνοβολομέλεια και συμμερίζομαι πολλές από τις απόψεις του. Η νέα έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα του HIV-AIDS μας αναγκάζει να τεθούμε σε επαγρύπνηση για το τι πρόοδο έχουμε επιτελέσει τα τελευταία 15 χρόνια. Παρόλα τα βήματα πρόοδου, μπορούμε να χάσουμε τα πάντα εάν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Ιδίως στο επίπεδο της πρόληψης. Ε, το ίμιση των φορέων του AIDS τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω έλλειψης θεραπείας και αγωγής. Από το 2011 βέβαια έχει εντατικοποιηθεί η πρόοδος, διότι τα αντίοικα έχουν πλέον χορηγηθεί σε πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS. Άρα έχει μειωθεί και σε σημαντικό μετραστικό τρόπο ο αριθμό των θανάτων. Όμω πρέπει να λάβουμε υπόψη και του κοινωνικού παράγοντε όπω τη φτώχεια, την ανισότητα και τις, τη διακρίση, τη διακριτική μεταχείριση. Ιδίω για του ευπαθεί πληθυσμού. Δηλαδή για αυτέ τι κατηγορίε ατόμων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν διακριτική μεταχείριση και να υποφέρουν από διακρίσεις. Κυρίως τα παιδιά. Έχουμε δει μεταξύ 2000 ε, και 2014 να μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που ε, μολύνονται, όμως ε, ακόμη ο αριθμός αυτός είναι ανησυχητικός ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα κατάλληλο εργαλείο κοινωνικής προστασίας που να επιτρέπει την πρόσβαση των μολυσμένων με τον ιό του AIDS στην ε, υγειονομική περίθαλψη για να λάβουν και την κατάλληλη αγωγή εγκαίρως. Ευχαριστούμε ο κύριος Γερέρος Αλόμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η διάσκεψη του ΟΗΕ θα λάβει γνώση των, ε, της πρόοδου που έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια σε αυτόν τον τομέα και στην πληροφόρηση η οποία βοηθάει στην πρόληψη ασθένειας ε, και στο ιατρικό και φαρμακευτικό τομέα ε, πιο μεγάλη δραστηριοποίηση της, κοινωνίας, των πολιτών ε, και υγειονομική περίθαλψη όλα αυτά μαζί και από κοινού κάνουν μια συλλογική προσπάθεια που προστατεύει πολλά εκατομμύρια ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Η πιο σημαντική όμως πρόοδος ε, που έχουμε πετύχει είναι η προσήλωση σε αυτόν τον αγώνα κατά της ασθένειας. Ακόμα 40 εκατομμύρια άτομα ε, ε, έχουν τον ιό του AIDS, πάνω από 2 εκατομμύρια πέθαναν το 2015 και συνεχίζουμε να βλέπουμε κρούσματα σε όλα, πολλά μέρη του κόσμου. Η Αφρική, η Ήπειρος του πόνου ε, και της φτώχειας εξακολουθεί να χάνει πολλούς ε, ανθρώπους της ε, εξαιτίας αυτής της ασθένειας. Σημαντικό είναι λοιπόν αυτή η δέσμευση και σε αυτή τη δέσμευση το πιο πάλι σημαντικό είναι τα 3-90%. 90% όσων έχουν τον ιό ε, να διαγνώσκονται από τα συστήματα. Το 90% αυτών που έχουν διαγνωστεί να λαμβάνουν αγωγή και το 90% όσων λαμβάνουν αγωγή να ε, ε, γλιτώνουν ε, και να θεραπεύονται. Αυτή θα πρέπει να είναι η στόχη μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να τα ενθαρρύνει να επεξεργαστούν συνολικά σχέδια τα οποία ε, θα περιλαμβάνουν και τη διάγνωση και τη θεραπεία αλλά και θα ε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα χωρίς διακρίσεις. Η Ισπανία έχει ε, εθνική στρατηγική αλλά έχει αποδυναμωθεί και αυτή τη στιγμή η η καταπολέμηση του AIDS δεν είναι αρκετή ε, διότι αυτή τη στιγμή αυξάνουν τα κρούσματα ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μειώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Συγκεράνης για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την δημόσια για το 2006, χωρίς αμφιβολία, είναι η διάσκεψη για την επαναχρηματοδότηση του Παγκοσμίου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS. Ένα καινούριο ραντεβού το οποίο προτίθεται σε αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Επιτροπό. Η διεθνή λοιπόν κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει τι ευθύνε τη, το να ε, σταματήσουμε να επαγρυπνούμε σε ό,τι αφορά τι απειλέ όχι μόνο του AIDS αλλά και άλλων ασθενειών όπω η ελανοσία και η φυματίωση. Θα σημαίνει να είμαστε με παροπίδες. Θα πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Ταμείο το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2002 θα πρέπει να ελπίζουμε ότι και η Κομισιόν αλλά και όλα τα κράτη-μέλη Όπω και το σύνολο των βιομηχανοποιημένων χωρών θα καταλάβει πόσο είναι σημαντικέ οι προτεραιότητε σε ό,τι αφορά την καθολική διάσταση τη παγκόσμια υγεία, Σε ό,τι αφορά το AIDS συγκεκριμένα, αυτοί που ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να αντιταχθούν στην ανάπτυξη θεραπείας, ε, στην πρόσβαση δηλαδή των ασθενών στα αντιϊκά, αυτοί αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι η στάση τους και η υπερβολή τους τότε ε, μας οδήγησε, θα μας είχε οδηγήσει σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Η πρόσβαση σε, για όλους ε, θα είναι... Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πραγματικότητα ε, για όλους σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα αυτά. Αυτό έχει τεθεί ως στόχο από το 2000. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τις ευθύνες της και τώρα λοιπόν στα κράτη-μέλη αφιέται να εφαρμόσουν αυτά που αποφασίστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάντσο έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, το HIV είναι πλέον παγκόσμια επιδημία. Μεταξύ του 1981 και του 2007 σκότωσε τουλάχιστον περίπου 25 εκατομμύρια άτομα και σήμερα πάνω από 30 εκατομμύρια άτομα έχουν μολυνθεί ε, ε, σε όλο τον κόσμο. Η Σύνοδος κορυφής, ε, υψηλού επίπεδου μάλλον του ΟΗΕ, ε, θα βοηθήσει να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά της επιδημίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει αυτό το θεσμό. Όχι όμως μόνο με λόγια για να είναι πραγματική αυτή η υποστηρίξη θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς αναπτύσσουμε ε, φάρμακα. Τα φάρμακα θα πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κόσμου και όχι των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Ε, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να επιτρέψουμε μέσω εμπορικών ε, συμφωνιών που θα περιλαμβάνουν διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας λέω να ευνοήσουμε την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα σε όλο τον κόσμο. τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα στο 95% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και αυτά τα λέει ο ΙΕ, όχι εγώ. Ο πιο κοινό τρόπο μόλυνση είναι, εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική μετάδοση. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προστασία παρόλο ότι ορισμένοι φανατικοί ε, δεν το δέχονται. Η καλύτερη προστασία είναι αυτό το προφυλακτικό. Και το είπε αυτό και το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προστατευτικά μέτρα όπω το προφυλακτικό ανδρικό και γυναικείο, καθώ επίση και να ενισχυθεί η αυτονομία των γυναικών στι σεξουαλικέ του σχέσει. Καλύτερη λοιπόν περισσότερη συνέπεια και περισσότερο ε, σεξ με πληροφόρηση και προστασία. Και κυρίω για τι γυναίκε. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Χάουταλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το γεγονός ότι στην Αφρική αυτή τη στιγμή μειώνονται τα κρούσματα του AIDS, τα νέα κρούσματα AIDS και όσοι ακολουθούν αγωγή δείχνουν ε, καλά αποτελέσματα αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσει που κάναμε στην πρόληψη για την ε, αναχέτηση του διάδοση του HIV μπορεί να μας αποδεχθεί πολύ ε, αποτελεσματική τεχνική μέχρι το 2020. Πρέπει λοιπόν αυτή τη δουλειά, την προληπτική, ε, καθώς και ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, να συνεχίσουμε τις σχετικές προσπάθειες, να τις εντατικοποιήσουμε. Χρειάζεται και μία ανάλογη πολιτική όχι μόνο για το AIDS αλλά και για τα φάρμακα που παρέχονται, για την πολιτική μας σχετικά με τα ναρκωτικά και τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ακόμα και για όσους προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Ευχαριστούμε ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, συνολικά ο στόχο μας είναι να αναχαιτήσουμε αυτήν την ε, επιδημία μέχρι το 2020, όμως να πετύχουμε ποτέ το στόχο αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Αφρική, ιδίω στην κεντρική και δυτική ε, Αφρική. Πρέπει να επιταχύνουμε την πρόσβαση στην αντιοική αγωγή για τους περισσότερους φορείς, διότι μόνο ένα τρίτο του πληθυσμού αυτή τη στιγμή έχει τέτοια πρόσβαση. Από τις 35 χώρες που συνεισφέρουν 90% ε, που έχουν μάλλον 90% των κρουσμάτων ε, στην ε, κατηργοποίηση του HIV AIDS παγκοσμίω, οι περισσότερες είναι αφρικανικές. Η, η Ιταλία είναι σε μια από τις πρώτες θέσεις έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια και το 2014 έχουμε 900.000 νέες ε, περιπτώσεις που διαγνώστηκαν του HIV. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε δραστικά μέτρα πρόληψης και να προβλέψουμε και νέες ε, δημοσιονομικές γραμμές για τις επενδύσεις. Πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται στι χώρε με μέσο και χαμηλό εισόδημα. Κάποιε φορέ μπορεί να φτάνει το 90% η τιμή των φαρμάκων σε σχέση με τη μέση παγκόσμια τιμή. Υπάρχει επίση τεράστια έλλειψη τέτοιων φαρμάκων στον δημόσιο τομέα, ενώ και ο ιδιωτικό τομέα έχει τεράστιε ανάγκε, αλλά οι τιμέ εκεί είναι και πολύ υψηλότερε. Αυτό λοιπόν επηρεάζει ιδιαίτερα τον πληθυσμό των φορέων. Υπάρχει πρόβλημα πρόσβαση στα φάρμακα, στην αγωγή στην Αφρική και ταυτόχρονα έχουμε πρόβλημα ε, υπέρ, υπέρμετρη προσφορά στι πλουσιότερε χώρε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη βιομηχανική παραγωγή των φαρμάκων, γιατί βρίσκεται στα χέρια λίγων φαρμακευτικών εταιριών που μπορούν να ορίζουν τι τιμέ και να, κανονίζουν τους, να ε, ρυθμίζουν του κανόνε ε, αντί να υπάρχουν πραγματικά έρευνες και να μην, να μην στοχεύουν μόνο στο κέρδος. Πρέπει λοιπόν να ε, ελέγξουμε κάπω τι κάνουν και αυτοί οι φαρμακευτικοί όμιλοι, γιατί πρόκειται για πραγματικό σκάνδαλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πίτικα είναι για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη δήλωση στην οποία προέβη. Κατέδειξε πραγματική δέσμευση. Δέσμευση προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα του AIDS και του HIV και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό στην Ευρώπη να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την πρόκληση αυτή. Η πρόκληση λοιπόν αυτή είναι τεράστια. Θα πρέπει όμως παράλληλα να θυμόμαστε ότι η καταπολέμηση, ο αγώνας κατά του AIDS, ε, HIV αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορεί να σταθεί με επιτυχία το θέμα της ε, διεθνούς συνεργασίας. Προωθούμε λοιπόν θέματα πρόληψης και αυτό καταφέραμε να το προωθήσουμε και έτσι στις περιπτώσεις αυτές ε, μπορούμε να βοηθήσουμε προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για, τους, για το θέμα που έχουν προσβληθεί. Ασφαλώς αυτό δεν αρκεί για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις μας συγκεκριμένα για να καταπολεμήσουμε το HIV έχουμε τέσσερις, ε, τέσσερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, χρειάζεται πρόληψη και η πρόληψη περιλαμβάνει και σεξουαλικά δικαιώματα για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι σχετίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζεται εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ο κόσμος ε, θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θεραπεία, σε αγωγή χωρίς να στιγματίζεται. Φυσικά εδώ το κλειδί είναι η πληροφόρηση. Και όπως γνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά συχνά συνδέονται και με θέματα κοινωνικού κύρους. Και θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Καμπέσον για ένα μισό λεπτό. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πάρα πολύ σημαντική και στην πρόληψη και στην ε, ε, θεραπεία του AIDS. Όμως ε, δεν μπορούμε να είμαστε πλέον ικανοποιημένοι διότι η πρόοδος που έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια κινδυνεύει αν δεν συνεχίσουμε και δεν ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ακόμα έχουμε 40, εκατομμύρια άτομα μολυσμένα, 22 εκατομμύρια από αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στην, σε αγωγή κατά του ιού. Ε, στην έκθεση μας για τα φάρμακα θα πρέπει εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το συμπεριλάβουμε καθώς επίσης και όλες τις πτυχές ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι αυτά τα άτομα πιο πολύ πλήττονται. Οπότε χρειάζεται να τονίσουμε και τη διάσταση του φύλου. Ε, στην Ευρώπη οι χώρες της ε, μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων έχουν αντιμετωπίσει ακόμα ακόμη πιο σοβαρά το πρόβλημα. Και θα ήθελα να ε, προειδοποιήσω διότι με την οικονομική κρίση και με την αλλαγή της χρήσης από κοκαίνη σε ηρωίνη που είναι πιο ε, φτηνή μπορεί να, δούμε στο μέλλον μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων AIDS ε, στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας με φιλόδοξου στόχους να εξαλείψουμε την επιδημία μέχρι το 2030. Χρειαζόμαστε εθνικά σχέδια ε, πρόληψης και θεραπείας και βέβαια να ενισχύσουμε τα συστήματα υγεία μας όπου θα πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση όλων, την καθολική πρόσβαση σε αυτά όλων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαρία για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, είναι προφανές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ιό του AIDS. 6 ε, εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη από αντιϊκά φάρμακα και έχουμε και ε, περισσότερα κρούσματα σε σχέση με το έτος 2000 τα τελευταία χρόνια. Φτάνουμε το 42% την ετήσια αύξηση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Αυτό που δεικνύουν οι μελέτε. Πρέπει να δώσουμε αξιοπρεπή συνθήκε ζωή σε όλου αυτού του φορεί. Δύο εκατομμύρια άτομα που ακόμη δεν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη αγωγή. Και δεν, ε, επίσης υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες, ε, κύριε, κυρίες και κύριοι, στον 21ο αιώνα. Ε, τέτοιες ε, αποκλήσεις, το τι πρόσβαση έχει ο ένας και ο άλλος ανάλογα με τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σφαιρική παγκόσμια στρατηγική ε, συντονισμένη, ώστε να υπάρξει κινητοποίηση, ε, χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις για τον αγώνα κατά του AIDS, ιδίω σε χώρε που έχουν περισσότερο ευπαθεί πληθυσμού ή περισσότερο ευπαθή συστήματα υγεία, αλλά και για τι ομάδε του πληθυσμού που είναι πιο εκτεθειμένε και προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πρόληψη στον αγώνα κατά του AIDS. Πρέπει να αφιερωσιώσουμε περισσότερου πόρου σε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να έχουμε έναν ενάρετο κύκλο σε αυτή την περίπτωση, μόνο εφόσον γίνουν οι κατάλληλε επενδύσει. Και γι' αυτό ελπίζουμε στη Σύνοδο του ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενώσει τι προσπάθειέ τη με του υπόλοιπου για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ευχαριστούμε κυρία Σένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμμετέχοντες ε, στην ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου θα πρέπει να λάβουν δεσμεύσεις προκειμένου ε, να, σταματήσει, να σταματήσουν οι διακρίσεις που υφίστανται οι φορείς του AIDS καθώς επίσης και να καταργήσουν τους νόμους που αυτή τη στιγμή ποινικοποιούν τους φορείς του AIDS σε πολλές χώρες. Θα πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα υγείας και αναπαραγωγικής υγείας και συνολικά. Ε, θα πρέπει να καταργηθεί το μονοπόλιο της ε, βιομηχανίας ε, και το, να λυθεί το πρόβλημα με, τις, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και τους εφήβους. Η έρευνα θα πρέπει να είναι δημόσια προς όφελος των πολιτών. Όχι να χρηματοδοτούμε με κρατικά χρήματα τις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες ε, που έχουν στο μυαλό τους μόνο το δικό τους συμφέρον και όχι το συμφέρον του λαού. Ευχαριστούμε κυρία Σένα. Δέχεστε μια γαλάζια καρτά από τον κύριο Αρνότ. Κύριε Αρνότ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι απλώς η εξής. Κατανοώ πλήρως το τι λέτε για τους φαρμακευτικούς ομίλους που ε, χρώνουν πολύ υψηλές τιμές για τα αντικά. Και καταλαβαίνω για ποιους λόγους λέτε ότι αυτό έχει αντίκτυπο στον αγώνα κατά του AIDS και του HIV. Η ερώτηση όμως είναι τι συγκεκριμένα θέλετε να κάνουν ε, τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτή τη συνάντηση υψηλού επίπεδου στο τέλος της εβδομάδας για το θέμα αυτό συγκεκριμένα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πιστεύω ότι το είπα σαφώς ε, στην παρέμβασή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση να ε, σταματήσει το εμπόριο των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να αποφασίσουν τα φάρμακα να πολλούνται σε οικονομικές χαμηλές τιμές. Ε, κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. 35 χρόνια φέτος κλείνουν από το πρώτο κρούσμα ε, AIDS, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την επιστημονική κοινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκέλος της έγκυρης διάγνωσης. Ακόμα πιο σημαντικό είναι η σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων. Η σωστή λοιπόν εκπαίδευση των νέων θα τους βοηθήσει να γίνουν υπεύθυνοι ενήλικες. Και σήμερα πιο πολύ από ποτέ είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υπεύθυνη συμπεριφορά γιατί βλέπουμε ανησυχητικέ τάσει βλέπουμε ότι είναι όλο μεγαλύτερος ο αριθμός παιδιών 10 έως 19 ετών που προσβάλλονται με HIV και έχουν χαθεί 30 εκατομμύρια ζωές από τον, τον ιό. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα έχει αποφανθεί ότι το 2, μέχρι το 2030 θα μπορούσαν να περιοριστούν δραματικά οι θάνατοι αν ξεκινούσε ε, άμεσα έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση αντιοικών. 22 εκατομμύρια άνθρωποι ακόμα δεν έχουν πρόσβαση σε αντιοικά και οι πιο πολλοί εξ αυτών δεν ξέρουν καν ότι έχουν μολυνθεί. Στην Υποσαχάρη Αφρική, σύμφωνα με μελέτες, 26 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φόρεις του HIV. Μεγάλος ρόλος λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, διάγνωση και την θεραπεία, την ε, χορήγηση αγωγής ε, είναι δραματίζεται από τι θρησκευτικέ κοινότητε σε ό,τι αφορά δηλαδή, την παροχή αγωγή Η κάρτα στην International πριν από δύο μήνε και άλλε θρησκευτικέ οργανώσει δημοσίευσαν κατευθυντήριε γραμμέ για την καταπολέμηση και την εκρίζωση των μολύνσεων μεταξύ των παιδιών μέχρι το 2020. Έχει πέσει αυτό το ποσοστό των παιδιών που μολύνονται και το 70% των γυναικών, των έγκυων γυναικών ε, που είναι φορείς του AIDS, του HIV, έχουν λάβει αγωγή προκειμένου να μην τα μεταδώσουν στα παιδιά τους. Η International Caritas και οι διεθνείς οργανώσεις, θρησκευτικές οργανώσεις εργάζονται προς την κατεύθυνση. Διακόπτει ο πρόεδρος, δυστυχώς. Και δίνει το λόγο στον κύριο Πόστ. Την κυρία Πόστ. Σας ευχαριστώ. Το κοινωνικό στίγμα και η διακριτική μεταχείριση είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την αγορά εργασία. Αυτό εξακολουθεί να οδηγεί σε μεγάλο ψυχικό, ψυχική επιβάρυνση για τα άτομα αυτά. Θα πρέπει να σταματήσει λοιπόν η στιγματοποίηση και θα πρέπει να υπάρχει επαρκή πληροφόρηση στην κοινωνία για την ασθένεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια κοινή απάντηση και όλοι να ταχθούμε υπέρ αυτή. Το μεγαλύτερο κίνδυνο για την διάδοση του AIDS είναι ακριβώς το στίγμα αυτό. Και το γεγονό ότι δεν αναζητεί το άτομο ενδεχομένω πληροφορίε και αγωγή όταν χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμούσουμε αυτό το στίγμα, την διακριτική μεταχείριση των μολυσμένων με HIV. Ο Η Παγκοσμία Οργάνωση Υγείας ε, τάσσεται υπέρ του αγώνα αυτού και χρειαζόμαστε προφανώς ε, πρωτοβουλίες και αρχές σε ευρωπαϊκό, κρατικό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά οργανώσεις οι οποίες θα αναλάβουν τα προγράμματα ενημέρωσης, προόληψης και υποστήριξης ασφαλώς και για τρίτα κράτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το και η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίτσα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η υποστήριξη της, ε, ε, των στόχων του ΟΗΕ για την εξάλληψη του ε, AIDS μέχρι το 2030 είναι και λόγος αλλά και ενθουσιασμός διότι στον Περμαίο, στο χωριό που γεννήθηκα το AIDS σκότωσε πάρα πολλά άτομα, υπερβολικά πολλά που εξαιτίας ε, της χρήση των ναρκωτικών ε, επλήγησαν και άρχισαν να πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο. Αλλά ταυτόχρονα ε, είδαμε και τις μητέρες, τις ε, οικογένειες ε, οι οποίες υπέφεραν πολύ και προσπάθησαν όμως και κέρδισαν αυτή τη μάχη. Αυτή τη ε, στιγμή ε, δεν πρέπει να χάσουμε αυτά που πετύχαμε ήδη. Το AIDS επιζεί ακόμα στο περιθώριο, στις ανισότητες, ε, στη φτώχεια, στις διακρίσεις και κυρίως έχει το πρόσωπο των γυναικών. Έχει σχέση με τον τρίτο κόσμο αλλά και με την Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να αποφύγουμε της, ε, την επιβολή των ακραίων απόψεων που υπάρχουν και αυτές. Το 2030 τουλάχιστον το 90% των φορέων θα πρέπει να το ξέρουν ότι είναι. Τουλάχιστον το 90% από αυτούς να λαμβάνουν αγωγή και τουλάχιστον το 90% αυτών που έλαβαν αγωγή να ε, θεραπεύονται στην πράξη από το AIDS. Ε, θέλουμε νόμους που δεν θα δυσκολεύουν την, την πρόσβαση. Θέλουμε περισσότερη ισότητα, ε, πιο συνειδητοποιημένες γυναίκες. Ε, ο στόχος είναι κοντά, μπορούμε να τον πετύχουμε. Ευχαριστούμε, αλλά υπήρξε μάλλον ένα πρόβλημα με τη διερμηνία στα γαλλικά. Κάποιοι συνάδελφοι δεν σας κατάλαβαν. Οπότε θα παρακαλούσα να τακτοποιηθεί αυτό. Όμως δεν μπορείτε να επαναλάβετε την ε, παρέμβασή σας. Παρακαλώ όμως ε, τις τεχνικές μας υπηρεσίες να το επιλύσουν. Επιλύθηκε τώρα. Α, ωραία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόλτσακ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για την πρόληψη. Κι άλλη πρόληψη χρειάζεται. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Ορθώς τονίζεται ο ρόλος που πρέπει να αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ταμείο για την καταπολέμηση της διάδοσης του ιού του AIDS και άλλων μεγάλων επιδημιών όπως η φυματίωση. Πρέπει να υπάρξει συσπηρωμένη ε, και συντονισμένη προσπάθεια από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου, η νόσος αυτή δείχνει πόσο η ιατρική αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Τη δεκαετία του 80 πρόκειται για μια αρρώστια ε, θανατηφόρα. Τώρα κάποιες φορές μπορεί και να θεραπευθεί ή τέλο πάντων να ελεγχθεί. Ε, πάντως είναι μια ασθένεια που κανείς μας δεν θέλει να έχει. Στην Ανατολική Ευρώπη ε, οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να φοβούνται, όμως τα 120.000 νέα κρούσματα ΥΟΣ δείχνουν ότι μάλλον τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Ο στόχο που είχαμε ε, θέσει ω το 2030, εκρίζωση, πλήρη εκρίζωση τη αρρώστιας, τη ασθένεια αυτή, είναι πολύ φιλόδοξος, Δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί. Περισσότερα λοιπόν πρέπει να επενδυθούν στην έρευνα και στην πρόληψη. Όπω είπαν αρκετοί από του συναδέλφου. Δυστυχώς η χώρα μου, η Δημοκρατία της Τσεχίας, επίσης δεν τα καταφέρνει καλύτερα σε αυτό το τομέα. Έχουμε ε, καταργήσει και ανακαλέσει κάποια προγράμματα πρόληψης που λειτουργούσαν ως τώρα και δυστυχώς αυτό έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από τότε που αρχίσαμε να συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς πρέπει να επενδύσει στην καταπολέμηση αυτής της ασθένειας, αλλά να επενδύσει και στην έρευνα και να στηρίξει τις χώρες που βρίσκονται στο άλλο μέρος της κλίμακας της στόχιας και δεν μπορούν να δώσουν φαρμακευτική αγωγή στους φορείς. Ευχαριστούμε. κυρία Σάλτε Μόζε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου είπατε ότι έχω 1,5 λεπτό. Ε, ωστόσο, ενώ έχω το λόγο, ε, να έχετε κατά νου ότι τρει άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή του λόγω του AIDS στον κόσμο. Ένα άνθρωπο πεθαίνει κάθε 30 δευτερόλεπτα. 40 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φορεί αυτή τη στιγμή. Και άλλα 2 εκατομμύρια προστίθενται ετησίω. Ε, είμαστε Τυχερή βέβαια, διότι υπάρχει και μια καλή είδηση. Έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε κάτι για το θέμα αυτό και να εκριζώσουμε την επιδημία του AIDS πριν από το 2030. Και γνωρίζουμε από τους στόχους της χιλιετίας και την αναθεώρηση της το 2015 ότι φέρνουν αποτελέσματα, διότι τουλάχιστον έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση στον αγώνα αυτό. Παρ' όλα αυτά μας ανησυχεί ε, έντονα να διαβάζουμε στην έκθεση του ΙΕ ότι εφόσον εξακολουθήσουμε να ενεργούμε όπως ως τώρα έχουμε κάνει με τα μέτρα που ως τώρα έχουμε αναλάβει περισσότερη φαίνεται τελικά οι του AIDS από ό,τι ε, επιδιώκαμε. Χρειάζεται λοιπόν εντονότερη δράση, περισσότερη χρηματοδότηση, πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί η φαρμακευτική αγωγή, διότι σε πολλές περιπτώσεις ενήλικοι στους οποίους χορηγείται η αγωγή δεν ε, καταφέρνουν τίποτα, δεν αντιμετωπίζουν την ασθένεια, διότι ε, μπορεί να μην έχουν τη σωστή συμπεριφορά. Ε, χρειάζεται λοιπόν και πολλή ενημέρωση. Δεν αρκεί απλώς να παίρνει κανείς φάρμακα όταν είναι φορέα. Θα πρέπει το AIDS να γίνει προτεραιότητά μας ε, και να το αντιμετωπίσουμε με ακόμη σοβαρότερο τρόπο. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Το 2000, μεταξύ 2009 και 2014 μειώθηκε κατά 45% ε, ο αριθμός των παιδιών που μολύνθηκαν με HIV. Η πρόληψη στις γυναίκες ε, και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες εξακολουθεί να αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση. Ένα πρόβλημα λοιπόν ε, έγκυται στο γεγονός ότι στις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση στην Αφρική, μόνο το ίμιση των παιδιών που εκτέθηκαν στο EOHIV πέρασαν από ιατρική εξέταση. Ένα τέταρτο της αγωγής λοιπόν για τον ιό του HIV, τον την φρουτσροντίδα στο δίνουν οι καθολικές οργανώσεις. Θεωρούν ότι αποτελεί του τους ευθύνη αυτό και για παράδειγμα, από την ε, Σλοβακικό Σχολείο της Αγίας Ελισάβετ στην ε, Σλοβακία χορηγείται βοήθεια σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τις μητέρες ε, της Αφρικής που μόλυνται με τον ιό. Σε ό,τι αφορά την άμβλωση ως λύση για κάθε πρόγραμμα υγείας θεωρούμε ότι σε ό,τι αφορά το παιδί, το παιδί για να γεννηθεί υγιές είναι φάρμακα της πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννησή του. Και οι εμπειρίες μας από την εργασία επιτόπου επιβεβαιώνουν ότι είναι πολύ σημαντικότερο να υπάρχει μια ίση σχέση μεταξύ των συζύγων παρά να υπάρχουν κλινικέ αμβλώσεων. Γιατί αυτή, αυτή η οικογένεια θα διδάξει και την ευθύνη στα παιδιά της. Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμε Επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όσα κάνει στο σκέλος της πρόληψης του AIDS και πραγματικά πολλά έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη έχουμε την καλύτερη ιατρική, την καλύτερη και πιο κορυφαία τεχνολογία ξέρουμε πώς να καταπολεμούμε την ασθένεια αυτή. Δυστυχώς τα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων είναι νέοι και αυτό πραγματικά είναι φρικτό. Μιλώ για τη χώρα μου, την Λετωνία. Και βλέπουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι η μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων είναι μεταξύ των νέων, γιατί χρησιμοποιούν νόμιμα α, ναρκωτικά, νόμιμες ναρκωτικές ε, ουσίες και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης με AIDS. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λοιπόν έχει χορηγήσει τρεις θεραπείες, τρεις αγωγές στην Λετωνία. Δυστυχώς τα κέντρα πρόληψης και τα μέτρα πρόληψης δεν διατίθενται προς όλους. Κυρίως σε άτομα που ζουν στην Ήπεθρο, στη χώρα μου και στο σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης ε, τα πράγματα είναι ασφαλώς πολύ καλύτερα από ότι ήταν στη δεκαετία του 90. Πολλοί από τους φορείς, από ό,τι βλέπουμε και από τα αριθμητικά στοιχεία, βρίσκονται στην υποσαχαρία Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και θρησκευτικέ ιδέες που προωθούν, για παράδειγμα, την σεξουαλική κακοποίηση, το οποίο προφανώς οδηγεί και σε ε, μόλυνση. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Καταρχάς, ο κύριος Χέι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω τον Επιτροπό εδώ σήμερα. Χαίρομαι για τη δουλειά που κάνει. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να συνεργαστούν εν ώψη αυτή τη συνάντηση υψηλού επίπεδου. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά ε, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικού υψηλού αριθμού ανθρώπων φορέων σε όλο τον κόσμο. 40 εκατομμύρια άτομα αυτή τη στιγμή είναι οι φορεί του έτσι σε όλο τον κόσμο. 16 εκατομμύρια τουλάχιστον ε, ζουν με το AIDS ε, λαμβάνοντας ε, θεραπεία, αγωγή. νομίζω ότι έχουμε φυσικάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο σε σχέση με το AIDS. Ε, στη δική μου χώρα πέρσι είχαμε τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων των τελευταίων πέντε ετών. και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι είναι φορείς. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και στην Ευρώπη πολλά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, στηρίζοντα ε, τη δράση του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το AIDS έχει οριστεί στην παγκόσμια ε, ημερήσια διάταξη και αφορά μια ολόκληρη γενιά. Τα πρώτα κρούσματα διαγνώστηκαν πριν από 30 χρόνια και το HIV έγινε σύντομα ένα παγκόσμιο δράμα. Αυτή τη στιγμή είναι εκατομμύρια οι φορεί που ζουν με τον ιό αυτό, ενώ λιγότερο από του μισού έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να έχουμε ε, συγκεκριμένου στόχου, αλλά αυτοί που ήδη έχουμε είναι πολύ φιλόδοξοι και σύντομα λέγει προθεσμία για την υλοποίησή του. Πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν με τη μείωση του αριθμού ε, των ε, φορέων και την πρόσβαση των φορέων στην φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μην συνεχίσει η μετάδοση του ιού αυτού. Πρέπει στη συνάντηση ψηλοπεπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να ληφθούν τολμηρέ αποφάσει που δεν αμφίσουν απ' έξω κανέναν, διότι ο αγώνα κατά του AIDS εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που θα εφαρμοστούν. Οι τεχνολογικέ και επιστημονικέ λύσει που έχουμε στη διάθεσή μα μπορούν να επιτρέψουν να επιτύχουμε του στόχου ε, τη ε, εκρίζωση τη νόσου μέχρι το 2030 μέσω του ΟΗΕ, αλλά μόνο εφόσον τα εργαλεία αυτά διατεθούν σε όλου και μπορέσουν να διατεθούν σε όλους το, με τον ίδιο τρόπο κυρίως στις στοχές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την επικείμενη συνάντηση εκπροσώπων των κυβερνήσεων και των δομών υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση του HIV, που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Ιουνίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών για το HIV είναι ιδιαίτερα ενισχυτικά, καθώς αποδεικνύεται ότι 36,9 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με τον ιό του HIV. Η Αφρική παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο της πανδημίας με 25,8 εκατομμύρια άτομα να είναι φορείς του AIDS το 2014. Παρά την μεγάλη αύξηση από το 2000 τη παγκόσμια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του, ο ιός του HIV-AIDS παραμένει αυξανόμενο με τέσσερα εκατομμύρια συνανθρώπου μα να έχουν προσβληθεί Αποδεικνύοντα ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση του hiv εξακολουθούν να είναι ανεπαρκεί. είναι επομένω αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να επενδύσει κονδύλια στην έρευνα για την παραγωγή ισχυρών και αποτελεσματικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του aids ενώ πρέπει να υπάρξει μέρημνα ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού παγκοσμίω να έχει πρόσβαση σε κατάλληλη ενημέρωση πρόληψη παροχή συμβουλών ιατρικών ελέγχων και θεραπεία για το aids. ευχαριστώ. θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, μια προσωπική μου εμπειρία ως παράδειγμα. Από την δεκαετία του 90 το παράδειγμα αυτό μου δίδαξε ότι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση είναι άκρο σημαντική και ότι όσοι είναι φορείς του AIDS μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κοινότητα όπου ζουν διότι έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, έχουν συζύγους που πρέπει να αντιμετωπίσουν τους γειτονές τους κάθε μέρα. Αυτά στη δεκαετία του 90 και αυτός ο γνωστός μου που είχε AIDS ζούσε σε μια πολύ μικρή πόλη. Θέλω να τονίσω το εξής. Η μόρφωση, η πρόληψη είναι ε, οι δύο τομεί στους οποίου πρέπει να επενδύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να έχει εδώ ηγετικό ρόλο. Μόνο εφόσον ευαισθητοποιούμε και ενημερώνουμε και είμαστε ανοιχτοί στις δημόσια συζητήσεις για το θέμα αυτό. Μόνο εφόσον επενδύουμε στην αγωγή, την εκπαίδευση και την πρόληψη μπορούμε να κρυζώσουμε αυτή την ασθένεια. Ευχαριστούμε και τώρα Επίτροπος κ. Ανδριουκάητη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τι προτάσει για ε, ε, προτάσεις ε, πρόορη διάγνωση, πρόσβαση σε όλους, εθνικές πολιτικές, την διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θέματα τιμολόγηση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, ιδιαίτερη προσθέση για τα παιδιά και ιδίως τα κορίτσια, ε, περισσότερες επενδύσεις ε, και τιμές οι οποίες ε, θα είναι αρκετά οικονομικές για να αυξηθεί η πρόσβαση. πολύ καλές όλες αυτές οι προτάσεις και η συνεισφορά σας. Είναι σαφές ότι η καταπολέμηση του AIDS δεν έχει ολοκληρωθεί παρόλες τις μεγάλες πρόοδους που έχουν σημειωθεί το AIDS επηρεάζει όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων που έχει κάθε χώρα να ανταποκριθεί. Το AIDS επίσης επηρεάζει τους πιο ευάλωτους και δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό το λόγο η αλληλεγγύη και η δράση μας θα πρέπει να είναι κοινή, συλλογική και προς όλους. Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να στηρίξουν την καθολική πρόσβαση σε αγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βοηθάει και τι γειτονικέ τη χώρες και όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Είμαι σίγουρο ότι η συνάντηση του υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ αργότερα αυτή τη βδομάδα θα στείλει ένα ε, ισχυρό και ενωμένο μήνυμα απόλυτη, και ενωτικό μήνυμα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.